El señor presidente. En Cerreruda eh, sesión. Ανανεώνεται η σύνοδο, συνεχίζεται η σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διακόπη προηγουμένω. εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσει, θεωρούμε ότι έχει εγκριθεί η μέση Το πρώτο σημείο είναι η σύσταση δεύτερης ανάγνωσης